Ε, Θέλω να σας πληροφορήσω καταρχήν κυρίες και κύριοι για την δύσκολη κατάσταση η οποία επικρατεί στην Πολωνία λόγω των τραγικών πλημμυρών στην Πολωνία. Ένα μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι αυτή τη στιγμή κάτω από το νερό και χάνουν τις περιουσίες τους και τη ζωή τους άτομα εκεί. Θέλω να εκφράσω λοιπόν την απόλυτη αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας στο λαό της Πολωνίας. Θέλω να εκφράσω την βαθιά μας συμπαράσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι πλήττονται από τις πλημμύρες σήμερα στην Πολωνία. Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego 16 czerwca odbędzie Στις 16 Ιουνίου στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα κάνουμε μια συζήτηση για το ζήτημα αυτό και είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει μια απάντηση στο θέμα αυτό και θα ανταποκριθεί στην ε, αίτηση της Πολωνίας για υποστήριξη. Έχουμε ένα ταμείο ελεγγύη το οποίο διαδραματίζει ένα μεγάλο ρόλο για να ανακουφίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τέτοιες φυσικές καταστροφές. Κυρίε και κύριοι, σήμερα το πρωί υπήρξε μια συνάντηση της συνέλευσης των Πρόεδρων των Πολιτικών Κομμάτων και μόνο πριν από 10 λεπτά τελείωσε αυτή η συζήτηση, αυτή η συνεδρίαση τη Συνόδου των Πρόεδρων. Συζητήσαμε τα θέματα τη οργάνωση των ψηφοφοριών σε σχέση με το ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Θα γνωρίζετε φυσικά ότι η στρατηγική αυτή έχει σαν στόχο να δημιουργήσει θέσει απασχόλησης και να δώσει ευμάρεια στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει φυσικά και τη σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην επόμενη δεκαετία. Αυτή η στρατηγική είναι κομβική για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική, αυτή την στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον περιγυρό της, γιατί μπορούμε να είμαστε ισχυροί στον έξω χώρο αν είμαστε εσωτερικά συνεκτικοί. Στο φως των συζητήσεων λοιπόν στη συνέλευση των Προέδρων, ακούσαμε απόψεις και υπέρ και κατά του να ψηφιστούν τα ψηφίσματα για την Ευρώπη 2020 σήμερα, γιατί οικοθενοείται ότι θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν να εγκριθούν αυτά τα ψηφίσματα για να έχουμε και διαπραγματεύσει με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη σημαντική στρατηγική. Ακούσαμε όμω και επιχειρήματα που τονίζουν ότι θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική από την πλευρά του Κοινοβουλίου, η οποία να υποστηρίζεται από μια ευρύτατη πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να έχουμε μια ικανότητα επιρροή για τα θέματα αυτά έναντι των άλλων θεσμικών οργάνων. Και επειδή υπάρχουν αμφιβολίε σε σχέση με τη δυνατότητα να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία σήμερα, ναι, μεν θα θέλαμε να έχουμε μια ταχεία διεκπαιδεύση του θέματο αυτού, αλλά απαιτείται και μια ισχυρή πλειοψηφία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο φω λοιπόν των συζητήσεων αυτών μεταξύ των ηγετών των πολιτικών ομάδων, εγώ αποφάσισα να υποβάλω στην Ολομέλεια μια πρόταση αναβολή τη ψηφοφορία για την ε, Ευρώπη 2020 βάσει του άρθρου 140 του κανονισμού μας. <clears throat> Σας τονίζω και πάλι ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Είμαστε εν γνώση του γεγονότος ότι χρειαζόμαστε ένα ψήφισμα το ταχύτερο δυνατό, αλλά πρέπει το ψήφισμα αυτό να έχει μια ευρεία πολιτική υποστήριξη. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα τα οποία διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να σας υποβάλω λοιπόν αυτή την πρόταση και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συζητήσουμε τη δυνατότητα αναβολής της ψήφισης του ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020. Καταρχήν θα πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ και μετά κατά αυτής της πρότασης. Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο υπέρ της αναβολής, ο κύριος Ντόλ. Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι και οι Ούγγροι φίλοι είναι στην ίδια κατάσταση με τους Πολωνούς σε επίπεδο ε, των προβλημάτων με τις πλημμύρες. Πρέπει λοιπόν και για τους Ούγκρους να σκεφτούμε αντίστοιχα. Θα συμφωνήσω μαζί σας για την παρουσίαση την οποία κάνατε. Σε μια περίοδο κρίσης θα πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να συνεργάζονται. Υπό το πνεύμα αυτής της συνεργασίας είχα προτείνει στην διάσκεψη των Προέδρων πριν από τη συνάντηση του Στρασβούργου τις διαφορές ε, οι οποίες υπάρχουν σχετικά ε, με το θέμα αυτό ας αναβάλουμε την ε, απόφαση για τον μήνα Ιούνιο. Βέβαια δεν υπήρξε πλειοψηφία στη διάσκεψη των Προέδρων και γι' αυτό προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε το συγκεκριμένο ψήφισμα. Χθε το μεσημέρι όμως μετά από συζητήσεις Είδαμε ότι υπήρχαν ορισμένα κενά βέβαια. Δεν λέω ότι τα πράγματα παρουσιαζόντουσαν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θέλω να υποτιμήσω όλους αυτούς που πήραν μέρος στην προετοιμασία της έκθεσης για το 2020. Αλλά παρόλα αυτά διαπιστώθηκαν ορισμένα προβλήματα. Και γι' αυτό κάποιοι αρχηγοί αντιπροσωπιών είπαν ότι θα ήταν καλύτερο να ψηφίσουμε το θέμα την επόμενη φορά, τον μήνα Ιούνιο, γιατί η κρίση προφανώς δεν θα έχει τελειώσει μέχρι τότε. Συζητήσαμε λοιπόν από κοινού και καταλήξαμε σε μια συμφωνία και οι αρχηγοί των μεγάλων πολιτικών ομάδων ζήτησαν την αναβολή της ψηφοφορίας για τον μήνα Ιούνιο. Ο Μάρτιν Σούλτς μου είπε όμως θέλω την πλειοψηφία της ε, ομάδας μου. Όλοι έχουν ανάγκη την πλειοψηφία της ομάδας τους. Εμείς δεν συζητήσαμε στη δική μου συνεδρίαση χθε το βράδυ τροπολογίες, δεν συζητήσαμε επί της ουσίας γιατί η πλειοψηφία ήθελε την αναβολή της συζήτησης και της ψηφοφορίας για κάτι το τόσο απαραίτητο για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και γι' αυτό λοιπόν μετά από τη συζήτηση αυτή έλαβα και μία επιστολή και από τον κύριο Φερχόστατ και ζητάμε απλά την αναβολή κατά τρεις εβδομάδες του θέματος αυτού κάτω από τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση έτσι ώστε να προσδώσουμε περισσότερες δυνάμεις επιρροή στο κοινοβούλιο μας για να δείξουμε ότι είμαστε άνδρες και γυναίκες πολιτικοί κύρια υπεύθυνοι. Σας ευχαριστώ τώρα κατά της πρότασης αυτής. κύριος Σούλτσα ήθελε τον λόγο. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφος Ντόλ στην αρχή της παρέμβασής του αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση και στην Ουγγαρία. Σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή και οι Σλοβάκοι συμπολίτε μας πλήττονται από τις πλημμύρες αυτές. Νομίζω ανεξαρτήτως λοιπόν σε ποια χώρα βρίσκεται κανείς στην Ουγγαρία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία. Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους πολίτες που πλήττονται Κύριε Πρόεδρε, ο Ιωζεφ Ντόλ και εσείς ο ίδιος περιγράψατε την κατάσταση την χτεσινή και στην διάσκεψη των ε, Προεδρών από πλευράς διαδικασίας δεν έχω να προσθέσω τίποτα αλλά εξ ονόματος των συναδέλφων Μπίσκι και Κον Μπεντίτ θα ήθελα να πω πως δεν συμφωνήσαμε εμείς και υπερψηφίσαμε την πρότασή σας ε, την σημερινή περί αναβολής γιατί θεωρούμε πως πρέπει και μπορούμε να ψηφίσουμε. Υπάρχει επιθυμία ευρύτατη επιθυμία να έχουμε ε, μια ευρεία πλειοψηφία για αυτό το ψήφισμα αυτό όμως τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες μέρες δεν είναι διαδικαστικά αλλά ουσιαστικά είναι ξεκάθαρο ζήσαμε πως από πράγματα τα οποία ε, ήταν αντικείμενο συμφωνίας τον Φεβρουάριο πλέον δεν αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας και δεν είναι περίεργο αυτό λόγω της κρίσης. Υπάρχουν λύσεις που κάποιοι θεωρούν καλές, που είναι δημοκρατικά νομοποιημένες, κάποιοι άλλοι θεωρούν κάποιες άλλες καλύτερες και νομίζω πως κάποια στιγμή θα πρέπει να λάβουμε σαφείς θέσεις. Εσείς έχετε σαφείς θέσεις, εμείς έχουμε σαφείς θέσεις. Προσπαθήσαμε να τις συμβιβάσουμε, δεν τα καταφέραμε. Τώρα θα πρέπει να βρούμε πλειοψηφία είτε για τη μία είτε για την άλλη θέση. Εάν έχουμε πλειοψηφία για την αναβολή, θέλω να πω ήδη από τώρα πως εμείς ως σοσιαλδημοκράτες οπωσδήποτε δεν θα αποκλείσουμε νέα διαπραγμάτευση, αλλά αφετηρία θα είναι το κείμενο που ε, καταθέσαμε από κοινού με τους πρασίνους συναδέλφους. Οπότε θεωρώ πως πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής του ψηφίσματος για το 2020. Σας ευχαριστώ. Ποιος είναι κατά. Dziękuję. Σας ευχαριστώ. Otwieram głosowanie. Głosowanie elektroniczne. Λοιπόν, θα γίνει μια ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχιτη ψηφοφορία. Czy wszyscy zagłosowali? Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Λοιπόν, η πρόταση αυτή εγκρίθηκε. Αναβάλλεται η ψηφοφορία για το ψήφισμα για το 2020. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντόλ και τον κύριο Σούλτς για το ότι επεσήμαναν το ότι η πλημμύρα πράγματι έχει επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σωστά λέτε πρέπει να ε, επιδείξουμε την αλληλεγγύη μας με όλες αυτές τις χώρες και τις πολίτες. Κύριε Μπεζίνα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, μία παρατήρηση η πλημμύρα στην Πολωνία ξεκίνησε από την Τσεχία και είχε προκαλέσει μεγάλες ζημιές. Και, και η Τσεχία είναι μέλος της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από την Πολωνία. Πράγματι αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς είπα και εγώ όταν ευχαρίστησα τους κυρίους Ντόλ και Σούλτς για την